Το το μεσημέρι. Επόμενο σημείο στην ημέρηση διάταξη. Έκθεση της Ανθέα Μάκιντάερ όσον αφορά το τομέα της καλλιεργίας των ε, κυπεστικών. Θα τη δώσω το λόγο για 4 λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα αυτή την έκθεση και ελπίζω τελικά να υποστηριχθεί ευρέως ε, η καλλιέργεια των αθέων είναι σημαντικό θέμα για την Ευρώπη και νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει τα μάλα και στην ευρωπαϊκή οικονομία και να τροφοδοτήσει και τον κόσμο σε μια περιοχή που όλοι προβληματιζόμαστε για την ασφάλεια των τροφίμων. Η καλλιέργεια λοιπόν, η φυτοκαλλιέργεια μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά τονίζει τη σημασία που έχει να προωθήσουμε την καλλιέργεια των κυπευτικών και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε καλύτερα στην παγκόσμια αγορά μέσω καινοτομία, μέσω έρευνα, ανάπτυξη, αποδοτική φύση τη ενεργεία, προσαρμογή στι αλλαγέ του κλίματο. Όλα αυτά καλύπτονται σαν στοιχεία στην έκθεση. Η ασφάλεια τη διατροφή των τροφίμων είναι σημαντικότατο θέμα, μα προβληματίζει όλου. Σε 20 χρόνια θα χρειαζόμαστε περίπου 40% περισσότερα τρόφιμα από αυτά που παράγουμε τώρα και σε αυτή τη φάση η παραγωγή κυπευτικών παράγει το 18% ε, των προϊόντων γεωργίας της Ευρώπης και χρησιμοποιεί μόλις το 3% της γης. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο πρόθεσης του τομέα. Χρειαζόμαστε επίσης να μπορούμε να εξάγουμε και η έκθεσή μου τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης πρόσβασης των παραγωγών μας στις αγορές των χωρών. Η αξία των διακοσμητικών φυτών είναι περίπου 1,9 δις το χρόνο σε αξία εξαγωγών. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω, αλλά δεν θα έχω το χρόνο να τα καλύψω όλα. Η έκθεση στηρίζει τις οργανώσεις των παραγωγών και όλος ιδιαίτερος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεώρηση του καθεστώτος οπορικευαστικών που ετοιμάζεται σε αυτή τη φάση να μας δώσει σαφείς και πρακτικούς κανόνες όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας για τα, για τα κυπευτικά και να μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες σε διάφορα κράτη-μέλη που ισχύουν διαφορετικές συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, επίσης κάποια προϊόντα δεν έχουν χάσει την αναγνώρισή τους διότι τελικά τα προϊόντα αυτά δεν συμμορφώνονται στον τρόπο με τον οποίο θέλει να παράγονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ε, χρειάζεται να είμαστε πιο θετικοί όσον αφορά την προσέγγιση μας προς παραγωγούς και τις οργανώσεις των παραγωγών. Άλλη πτυχή είναι ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοπαρασίτων ε, είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο περιθώριο για μελλοντική ανάπτυξη αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε σε μια παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να ενστερνιστούμε νέες μεθόδους, νέες τεχνικές. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να διατηνόμεθα ότι απλώς θέλουμε να επιστρέψουμε στην βιολογική πράσινη καλλιέργεια, όπου δεν αγγίζουμε τίποτα. Αυτές οι μέθοδοι μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούμε τα προϊόντα, αλλά για την ώρα δεν μπορούμε χωρίς να έχουμε προϊόντα προστασία των φυτών, διάφορα είδη ψεκασμού και νεοκτενοειδή. οποιουσδήποτε αποφάσεις θα λάβουμε πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και όχι απλώς σε αντιμετώπιση των εμφανιζομένων κινδύνων. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στις οργανώσεις όπως το Πανεπιστήμιο του Harper Adams, τα Δυτικά Midlands, ε, που έχουν δραστηριοποιηθεί πολύ τα πανεπιστήμια σε αυτό το τομέα βλέποντας τα επίπεδα της ενεργείας των νέων σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες να προσφέρουμε καριέρες που αξίζουν τον κόπο στην παραγωγή, τον κυπευτικό. Χρειαζόμαστε βοτανολόγους, χρειαζόμαστε ε, ειδικού για τα φυτά, γεωπόνους. Και είναι καριέρες που αξίζουν τον κόπο και πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να προχωρήσουν προς αυτές τις κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάκιντάρ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα ας πάμε στη δικασία Catch